Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, ε, άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξης είναι η έκθεση Χάφνε σχετικά με την ε, σύναψη διοργανωτικής συμφωνίας και το χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου και δίνω αμέσω ε, το λόγο στον, στον εισηγητή κύριο Χάφνερ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ε, την ε, επίτευξη δημοκρατία στην Ευρώπη διότι η δημοκρατία βασίζεται στην ιδέα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κρυφά και ότι χρειάζεται διαφάνεια πρόσβαση του κοινού και οι πολίτες όπως και οι εκπρόσωποι τους οι εκλεγμένοι βουλευτές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται ή στην, ε, στον πολιτικό τομέα. Ε, αυτό μας έχετε ζητήσει μέσω των εκλογών σαν πολίτες. Οπότε <clears throat> σύμφωνα με τη νέα συνθήκη το Κοινοβούλιο έχει και τη δυνατότητα και την υποχρέωση να παρακολουθεί και την πολιτική και τις διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με την σύναψη νέων συμφωνιών για να μπορεί να τις και σήμερα δυστυχώς ε, έχουμε λήψει στο θέμα της μετάδοσης των πληροφοριών και στις συζητήσεις ε, ακόμη και ε, με το κοινό στο θέμα παραδείγματος χάρη της άκτα που έπρεπε να διαπραγματευτούμε συμφωνίες χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία και χωρίς να μπορούμε να κρίνουμε τι έχει συμφωνηθεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει και προφανώς θα αλλάξει μετά από αυτή τη συμφωνία την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνάψει ε, κατόπιν συζητήσεων με την Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τρόπον ώστε να έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα. Και εδώ δεν πρόκειται ε, μόνο σχετικά με τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων για ε, συνθήκες οι οποίες έχουν συναυθεί αλλά και για τον προγραμματισμό, τα εσωτερικά εμπιστευτικά απόρριτα και άκρος απόρριτα έγγραφα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία διαβαθμισμένη διαδικασία για το πόσο θα διεκπεραιώνουμε τα έγγραφα αυτά. Ε, πρέπει όμως όλα τα εμπιστευτικά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη διαβάθμιση να μπορούν να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ευρωβουλευτές. Βέβαια για τα άκρος χρειάζεται μια ειδική διαδικασία. Και θέλω να πω ένα πράγμα στους συναδέλφους. Η γνώση είναι δύναμη και εξουσία και πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε το Συμβούλιο. Αλλά θα πρέπει υπεύθυνα να ε, χειριστούμε τις γνώσεις που θα έχουμε αποκτήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν όλα τα οποία μαθαίνουμε να τα μεταδίδουμε προς τα έξω. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι Είναι όμως ένα βασικό βήμα για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ε, δημοκρατίας όχι μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ε, και του Συμβουλίου για να μπορούμε να έχουμε ε, πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Θέλουμε να ξέρουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ, στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ποιες είναι οι γραμμές γραμμές των διαπραγματεύσεων ποια είναι η διαπραγματευτική στρατηγική και ε, τι ακόμη το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, επιτροπές ε, ερεύνης που μπορεί να υπάρξει διαφθορά και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη. Δηλαδή δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα δεν μπορούμε να θίξουμε ορισμένους μάρτυρες και αυτό εν ονόματι της δημοκρατίας δεν είναι σκόπιμο. Διαφορετικά δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τους πολίτες εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και εύχομαι η συζήτηση να έχει ένα αίσιον πέρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα οι αγορητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ο κύριο Τρασκόφσκι. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τη διαπραγματευτική ομάδα και τον κύριο Χεύνα, τον επικεφαλής διότι πέτυχαν μια πολύ σημαντική συμφωνία Κάτι το οποίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ιδίω όταν εμπλέκονται δύο θεσμικά όργανα και όταν στο ένα ε, δίνονται νέε εξουσίε, ιδίω σε τόσο λεπτού τομεί, ευαίσθητου τομεί όπω είναι οι διαβαθμισμένε πληροφορίε. Στην προκειμένη περίπτωση, οι διαπραγματευτέ μα κατάφεραν να, ε, να πετύχουν μια πολύ όρημη συμφωνία, η οποία μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε διαβαθμισμένε πληροφορίε του Συμβουλίου. Σε πολλού μπορεί να φαίνεται τεχνικό το ζήτημα Πρόκειται όμως για ένα ακόμα βήμα προς την πρακτική υλοποίηση, κάτι που ακούμε εδώ, για κάτι που ακούμε εδώ και χρόνια. Ε, μετά δηλαδή από την έκκλησή μας για μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο αυτών που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τη διαφάνεια που αποτελεί προτεραιότητα για το κοινοβουλίο μας τα πολλά τελευταία χρόνια μετά τις αλλαγές ε, των συνθήκων. Θέλουμε να έχουμε την πιο πλήρη δυνατή εικόνα για να μπορούμε να αποφασίσουμε με τα λόγου ω κοινοβούλιο. Και όπω είπε ο κύριο Χέφνερ, όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία. Έχουμε τι εξεταστικέ επιτροπέ, την πρόσβαση πληροφοριών στου τομεί που διαπραγματευθήκαμε ή στον τομέα τη κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλεια που έχουμε ακόμη μπροστά μα. Η διαπραγματευτική μα ομάδα τα κατάφερε πολύ καλά το νομικό πλαίσιο, οι αρχές πλέον υπάρχουν και άρα επιτακτική ανάγκη πλέον είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να επιτελέσει το δικό του έργο και να θεσπίσει ένα σύστημα για να μπορούν αυτές οι συμφωνίες να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια ερμηνείας και ελπίζω το Συμβούλιο να συνεχίσει να επιδεικνύει ε, θετικό πνεύμα, πνεύμα συνεργασίας. Γνωρίζουμε ότι η ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατοχυρώνεται στις συνθήκες, αλλά είναι πολύ καλό να το βλέπει κανείς να παίρνει σάρκα και οστά. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον αυτό έγινε. Ιδίω δε όταν ξέρουμε ότι λείπει ένα ακόμη κομμάτι του πάζλ σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική εποπτεία και τον, ε, την πρόσβαση των, ε, του Κοινοβουλίου στα διαφασμισμένα έγγραφα της ΚΕΠΑ. Παραλαμβάνω ακόμα αυτό δεν έχει ακόμη επιληθεί. Επίσης ε, με τη βοήθεια της Οργανικής Συμφωνίας μπορούμε και εμείς να φέρουμε σε πέρα τα καθήκοντά μα στο Κοινοβούλιο καλύτερα έχοντας ενημέρωση και μπορώντας να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η προτεραιότητά μας άλλωστε, ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, του Συμβουλίου και αυτό το πετύχαμε και με τις αλλαγές των συνθηκών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Γκερέρος Αλόμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον κύριο Χέφνερ για την έκθεση που συζητούμε σήμερα και την οποία εν συνεχεία θα ψηφίσουμε. Αν δει κανεί ε, τα δημοκρατικά εγχειρίδια ή οι ειδικέ ε, μελέτες ε, θα δούμε διάφορους ορισμού για το τι είναι η δημοκρατία. Αλλά στις αρχές του 21ου αιώνα δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ένα καθεστώ της κοινή γνώμης και της διαφάνειας, της δημόσιας κοινή γνώμης. Οι θύνοντες δεν είναι μόνο ε, υπόλογοι απέναντι στην κοινή γνώμη και απέναντι στους αλλά θα πρέπει και να λογοδοτούν ε, σε σχέση με αυτά που πράττουν. Για να μπορέσουμε λοιπόν να φέρουμε σε πέρα στα βασικά μας καθήκοντα που είναι η νομοθέτηση και ο έλεγχος των ηθινόντων χρειαζόμαστε ενημέρωση, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Μόνο έτσι μπορεί το Κοινοβούλιο να φέρει σε πέρα την υποχρέωση που έχει να εκπροσωπεί του πολίτε που το έχουν εκλέξει. Τρία σημεία έχει η έκθεση που συζητούμε σήμερα. Θέλω να τα τονίσω αυτά. Πρώτα απ' όλα αυξάνει την αξιοπρέπεια των Ευρωβουλευτών, διότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου. Επίση, διευρύνει ε, τον αριθμό των βουλευτών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στι στις πληροφορίες, οι κοιόδης συγητέ, μέλη των ενδιαφερομένων επιτροπών και τέλος μειώνει ε, το πεδίο των διαπαθμισμένων πληροφοριών για τις οποίες ο βουλευτής ε, απαιτεί κάποιο είδους έγκριση, αδειοδότηση. Πρόκειται λοιπόν για ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός. Όπως ε, υπόθηκε, το μόνο που απομένει να δούμε τη διαδικασία που θα υιοθετήσουμε ώστε να μπορούμε με πιο οργανωμένο τρόπο να αξιοποιούμε αυτές τις διαβασμένες πληροφορίες και να λυθεί και το ζήτημα με τις διαβασμένες πληροφορίες της ΚΕΠΑ. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα σκόπελο στις ε, διαπραγματεύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τη διαπραγματευτική ομάδα, την κυρία Χάμς, την κυρία Βόλης, τον κύριο Λένε, τον κύριο Σβόποντερ που αρχικά ε, μας εκπροσώπησαν σε αυτή τη ε, διαπραγμάτευση. Κύριε Ρούμπιχ, ζητήσατε με την γαλάζια κάρτα να παρέμβετε. Δέχεστε, κύριε Γκερέρο, την γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ. <clears throat> Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν κάνει μία διαφορά σχετικά με τα απόρριτα του Συμβουλίου και από την άλλη πλευρά τα απόρριτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο πώς αξιολογεί τα δύο θεσμικά όργανα ή θεωρεί ότι και τα δύο είναι ισότιμα. Ουσιαστικά αυτή η συμφωνία αυτό που κάνει είναι ότι περιορίζει ε, το πεδίο των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Δεν το περιορίζει συνολικά, απλά δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα χωρίς καμία έγκριση ε, ασφαλείας, πρόσβαση σε αυτές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες πληροφορίες, φυσικά και πρέπει να είναι πιο ανοιχτή η ρύθμιση σχετικά το Κοινοβούλιο σε σχέση με τον αστραδιωτικό τομέα, όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, των προσώπων θα πρέπει να συνδέεται με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες αυτές. Ωραία. Και τώρα για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Γιατερμάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Χέφνερ για την καλή συνεργασία. Όπως και... Ευχαριστώ τον κύριο Χέφνερ. Έχουμε την ίδια άποψη. Χρειάζεται διαφάνεια και θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε. Πράγμα το οποίο ισχύει και για μας. Χωρίς πληροφορίες δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε ούτε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Εξού και τώρα πρέπει κάπου να καταλήξουμε ε, τώρα σχετικά με τις απαιτήσει διαφάνειας διαφάνειες οι οποίες υπάρχουν. δεν είναι ε, ίσως ένα τεράστι, μια τεράστια πρόοδος αλλά ε, ε, πολλές πληροφορίες ακόμη δεν καλύπτονται και δεν είναι δυνατόν οι πληροφορίες του PSP να είναι ε, ε, απόρριτες ε, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τα δίκτυα θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις για τα θεσμικά όργανα για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Φόξο για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω ε, καταρχήν τον κύριο Χάφνερ για την εργασία του σαν εισηγητή και η ομάδα μου συμφωνεί με αυτή την συμφωνία. Είναι σημαντική η εργασία για να μπορούμε να ε, ε, θεωρούμε υπόλογου στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δαπανούνται σωστά τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και ότι υπάρχει διαφάνεια και θεωρώ ότι η ρύθμιση αυτή με το Συμβούλιο ακολουθεί το πνεύμα της ρυθμίσεως που έχει επιτευχθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χαιρετίζω και καλύπτει και τον εμπιστοευτικό χαρακτήρα ορισμένων εγγράφων. Οπότε στηρίζω την έκθεση και πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε μια καλύτερη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο ε, στην κυρία Βερζιά θα έπρεπε να της δώσω το λόγο δεν τη βλέπω όμως μέσα στην αίθουσα και στον κύριο Αγκουράκη ο οποίος όμως δυστυχώς δεν είναι ακόμη στην αίθουσα ως εκ τούτου θα δώσω τον ε, λόγο σε όποιον τη ζητήσει με τη διαδικασία Catch the Eye και πρώτος είναι ο κύριος Έρενχάουζερ ίσως ε, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Έχουμε κάνει ορισμένες κοινοβουλευτικές επερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και υπάρχει και μια γραπτή επερώτηση εις ε, τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αριθμό των διαβαθμισμένων ε, εγγράφων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή δεν μας έδωσε απάντηση μας είπε ότι το διοικητικό κόστος θα ήταν πολύ υψηλό και ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει τον αριθμό των διαβαθμισμένων εγγράφων στο Συμβούλιο. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Μας είπαν πόσες ε, βαθμίδες διαβάθμισης υπάρχουν, πόσα διαβαθμισμένα έγγραφα έχουν ε, ε, υπάρξει και του συγχαίρω. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμη πρέπει να εξετάσουμε και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου η απάντηση ήταν ότι ε, πέρυσι ε, εστάλθηκαν 10 διαβασμισμένα έγγραφα ενώ βλέπουμε κάθε χρόνο πάνω από 10.000 έγγραφα διαβαθμισμένα στο διαδίκτυο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε πολλά διαβαθμισμένα έγγραφα δεν ε, έχουν ληφθεί υπόψη και αυτό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε σωστά την κοινοβουλευτική μας ε, εργασία ελέγχου. Όσο αναφορά τα διαβαθμισμένα έγγραφα θα πρέπει κανείς να δει και στις διάφορες ιστοσελίδες αν ο αριθμός αυτός αυξάνεται ή όχι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο μιλητής και εισηγητής κύριος Χάφνερ για δύο λεπτά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση, διότι εδώ δεν, δεν δρούμε για λογαριασμό μας, εκπροσωπούμε όμως τους πολίτες της Ευρώπης και έχουμε ένα βαρύ έργο, είμαστε να, υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της δημοσιονομικής ευθύνης μας έχουμε και νομοθετική ευθύνη και αυτή μπορεί μπορεί όντως να εξασκηθεί μόνο ε, αν γνωρίζουμε περί τίνος ομιλούμε διότι δεν είναι δυνατό στην πολιτική μία χείρα να μην ξέρει τι κάνει η άλλη. Στην πολιτική λέγεται ότι τα βασικά παραμένουν και καλυμμένα, δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες και ελπίζουμε ότι σήμερα με την ψηφοφορία θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε συνάψει μία συμφωνία αλλά η πρακτική μίας επικοδομητικής συνεργασίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Ελπίζω όμως ότι ασχέτως του εάν δεν λάβουμε αμέσως όλα τα έγγραφα ξέρουμε ότι χωρίς αυτή τη συνθήκη πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα δεν θα μας δίδοντο και δεν είναι δυνατόν ε, όταν συζητάμε παραδείγματο χάρη μία συνθήκη σαν την άκτα να διαπραγματευόμαστε χωρίς να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα έγγραφα ή στις συνθήκες με την ε, ε, Κίνα. Η συνάδελφος Χαούταλα έπρεπε επανειλημμένος να πάει στο Συμβούλιο και σαν πρόεδρος Επιτροπής μπορούσε να δει ορισμένα έγγραφα τα οποία όμως δεν ήταν προσβάσιμα για τον εισηγητή και νομίζω ότι η διαφάνεια είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν θετικά αυτό το νέο δικαίωμα και ευχαριστώ όλους ε, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου όπως άλλωστε και από πλευράς του Κοινοβουλίου τον κύριο Λένη, την κυρία Χάρντς, ε, την κυρία Γουόλης και τον κύριο Σόμποντα. Ευχαριστώ, έληξε συνεδρίαση και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση Γκέριγκερ για τις επιτρεπόμενες